διαφόρων εκθέσεων. Καταρχάς την έκθεση της κυρίας Αρενά «Φτώχεια, μια προοπτική με γνώμονα το φύλλο». Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελικώς αυτές οι δύο συζητήσεις οι οποίες ε, έχουν οργανωθεί μια μετά την άλλη αγγίζουν το θέμα της φτώχειας. Ε, ασχοληθήκαμε με την αριακή ένδυα. Τώρα κοιτάζουμε την ένδυα από, τον, από την προοπτική, από τη σκοπιά του φύλου. Τι συμβαίνει με τα φύλλα ε, στην Ευρώπη. Σήμερα πάνω από 64 εκατομμύρια γυναίκε ζουν σε κατάσταση συνθήκε φτώχεια. 48% από αυτέ είναι μόνε και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες τους. Θεωρούνται μάλιστα ευπαθέστερο κοινό προς την ε, φτώχεια. Οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι επικεφαλής νοικοκυριού, συνήθως πιο συχνά από άντρες και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε συνθήκες ένδυας και κοινωνικού αποκλεισμού με ένα φαύλο κύκλο φτώχεια για αυτές, τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Σήμερα 27% των παιδιών στην Ευρώπη ζουν με τον κίνδυνο να περάσουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας 20 εκατομμύρια παιδιά σήμερα σε συνθήκες φτώχειας. Επίσης είδαμε ότι τα μέτρα λιτότητας που συχνά είναι τυφλά και έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν απλώς επιδεινώσει αυτές τις ανισότητες και τον κίνδυνο αποδυνάμωσης των γυναικών και των παιδιών τους. Οι μεστολογικές αποκλήσεις συνεχίζουν σήμερα. Το ίδιο και των φτωχών εργαζομένων με επισφαλή καθεστώτα απασχόλησης και βεβαίως και τα συνταξιδοτικά προβλήματα. 39% απόκληση χάσμα στο επίπεδο των συντάξεων. Δηλαδή κίνδυνος φτωχοποίησης για τα άτομα αυτά, τις γυναίκες που είναι πιο ηλικιωμένες. Περιτώ να θυμίσω ότι ο στόχος της στρατηγικής 2020 προβλέπει μείωση 20 εκατομμυρίων των ε, ατόμων που κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το στόχο σήμερα. Πρέπει να διακόψουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Είναι 127 εκατομμύρια τα άτομα σήμερα στην Ευρώπη, 22 εκατομμύρια παιδιά και όλος ιδιαιτέρως στις ενηλίκους, Γυναίκε πλήττονται ιδιαίτερω από αυτό το φαύλο κύκλο. Έχουμε καθορίσει μια σειρά από συστάσει ώστε αυτό ο κύκλο φτώχεια επιτέλου να πάυσει. Η πρώτη μα σύσταση ζητά να εξασφαλίσουμε δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και την δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το υγειονομικό σύστημα και τη δικαιοσύνη. Πράγματι, ε, φαίνεται ότι όταν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι καλής ποιότητας και είναι μια πρώτη ε, γραμμή στην οποία έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι αυτοί, υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη κατανομή του πλούτου. Αυτό είναι ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας της κοινωνίας από τη φτώχεια. Δεύτερη σύσταση, η καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης στο της απασχόλησης, που μπορεί να προκαλούν να είναι πηγή φτώχειας για τις γυναίκες. Χρειάζεται συντονισμό των γονεϊκών αδειών, των αδειών μητρότητας, και των γονεϊκών γενικότερα επιδομάτων, ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα, τις καταστάσεις καθώ ε, καθώς και τα επισφαλή τα απασχόληση για τις γυναίκες. Τρίτη σύσταση. Είναι σημαντικό το ελάχιστο, ο ελάχιστο μισθός, η ελάχιστη αμοιβή στην καταπολέμηση της φτώχειας. Σήμερα στην έκθεση δεν ζητάμε έναν ελάχιστο μισθό, κάτι που θα ήταν πολύ να γινόταν, αλλά ε, ζητούμε να υπάρχει τουλάχιστον αναθεώρηση του συστήματος των ελάχιστων αμοιβών σε όλη την Ευρώπη και ανταλλαγή των των πρακτικών μέσα στα πλαίσια τη καταπολέμηση τη φτώχεια. Τέταρτη διεκδίκηση ε, όσο χειρότερα γνωρίζουμε το φαινόμενο, τόσο λιγότερο μπορούμε να του εξεύρουμε λύσει. Χρειαζόμαστε αξιοπιστότερα στατιστικά στοιχεία για την καταπολέμηση τη φτώχεια σήμερα στην Ευρώπη. Επίση, θέλουμε ένα σύστημα ε, ε, προστασία για τα παιδιά, όπω έγινε στην περίπτωση τη εγγύηση για του νέου. Υπάρχουν ιστίε φτώχεια, πολύ δραστήριε σήμερα στην Ευρώπη. Πρέπει να τι καταπολεμήσουμε με συγκεκριμένε δράσει, Να πλήξουμε συγκεκριμένα την φτώχεια των παιδιών ως φαινόμενο. Επίσης ζητούμε, και αυτό συντονίζεται και με την έκθεση που συζητήθηκε αμέσως προηγουμένως, κοινωνικές ε, τιμές ε, για την ε, πρόσβαση στην ενέργεια, για την πρόσβαση στο νερό, ε, να μην πέφτει κανεί στην παγίδα της φτώχειας και επίσης ζητούμε φορολογικές πολιτικές οι οποίες να παροτρύνουν ε, όλους να καταπολέμουν τη φτώχεια. Σας ευχαριστώ όλους και όλες, όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης προκειμένου να συντάξουμε και αυτές τις συστάσεις. Ε, ελπίζω να υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία και θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα στην Επιτροπή για τα θέματα της απασχόλησης που μας ταλανίζουν. Σας ευχαριστούμε. Η κατάσταση είναι όντω ε, περίπλοκη και δύσκολη. Όμως με τις σύντομες αυτές παρουσιάσεις περνάμε απευθείας στην διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Και τώρα έχουν ζητήσει υπερβολικά πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Ας ε, κάνουμε το εξής λοιπόν. Θα δίνω το λόγο σε όσους πρόλαβαν να εγγραφούν εγκαίρως στον κατάλογο αγορητών. και όσοι έχουν ήδη μιλήσει σήμερα το απόγευμα μέσω της διαδικασίας ΚΑΤΣΔΙΑΗ δεν θα πάρουν ξανά το λόγο. Η κυρία Σόιντρο. Ε, πρόεδρε, η έκθεση αυτή περιέχει σημαντικά δεδομένα που ξεκαθαρίζουν ότι ακόμα και στις ευρωπαϊκές ε, κοινωνίες ε, περισσότερες γυναίκες κινδυνεύουν από φτώχεια από ότι άντρε, Η έκθεση λέει πως ο λόγος είναι η διακρίση στην αγορά εργασία και στις αμοιβέ. Είναι η, έξι, η έκτη έκθεση το 2016 που έχει παρόμοιο θέμα. Και δυστυχώ κατά την απόψή μου, δεν προτείνει κάποια καινούργια λύση. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική διακριτική μεταχείριση. Οι γονεί, παραδείγματο χάρη, υφίστανται διακριτική μεταχείριση γιατί ασχολούνται με τα παιδιά τους και δεν δουλεύουν. Θεωρώ πως ε, οι μητέρες και οι πατεράδες που ασχολούνται με τα παιδιά τους ε, υφίστανται διακριτική μεταχείριση γιατί η κοινωνία δεν το ανταμείβει. Και όσο ισχύει αυτό, οι γυναίκες θα υφίστανται και αυτές ε, διακριτική μεταχείριση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή είναι πραγματικά σκληρή και τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες υποφέρουν, υφίστανται διακρίσεις και βεβαίως ε, Γι' αυτό στο παρελθόν είχαμε αναλάβει κάποιες ε, πρωτοβουλίες για να είναι σε καλύτερη κατάσταση οι γυναίκες όταν είναι παραδείγματο χάρη θύματα εγκλημάτων. Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα πρέπει να είναι αυτόματο κάτι τέτοιο και το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στον κοινωνικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιούρακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ένδια είναι μια κατάσταση που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Το γνωρίζουμε πολύ καλά στην Πολωνία γιατί αυτή τη στιγμή θεσπίζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες που θα βελτιώσει την κατάστασή τους. Δεν κατανοώ γιατί στην έκθεση αυτή η άκρα αριστερά έχει περιλάβει στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της αντιμετώπισης της ένδυας των γυναικών. Γιατί ζητούμε να υπάρξει ε, αναγνώριση των οικογενειών ΛΟΑ. Τι είναι μια οικογένεια μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι φαινόμενα αυτά τα οποία αναγνωρίζονται. Δεν είναι θέμα της ένδυας για τις γυναίκες ή η δυνατότητα να έχουν όλοι το δικαίωμα να παντρευτούν άτομα οποιοδήποτε φίλου. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τον κόσμο στον οποίο έχουμε κατακτήσει την ελευθερία μέσα. Η κυρία Μπιλμπάου Παραντίκα έχει το λόγο. <coughs> Χωρίς μικρόφωνο. Η Ευρώπη στην Ευρώπη εξακολουθεί να έχει το γυναικείο πρόσωπο Έχουμε όλο και μεγαλύτερη δυσκολία ως γυναίκες να έχουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουμε λιγότερες αμοιβέ και αυτό φαίνεται και στις ε, συντάξεις μας. Αναλαμβάνουμε τη, τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα στο σπίτι. Και αυτό δεν γίνεται γιατί έχουμε λιγότερα προσόντα ή ικανότητες. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές για να δώσουν σε όλες τις γυναίκες στην Ευρώπη ένα ε, εισόδημα το οποίο θα είναι αξιοπρεπές και την πρόσβαση στην παιδεία και την κατάτηση. Πρέπει να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία των γυναικών, καλύτερη είναι και η δυνατότητα να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Οι περικοπές της λιτότητας όμως έχουν εμποδίσει τα προγράμματα αυτά, τα οποία είναι μια πραγματική επένδυση στο μέλλον. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική επανάσταση στη χώρα των ε, Βάσκων, που είναι η πέμπτη χώρα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, έχουμε ήδη επιτύχει να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά μόνο να υποστεί τι συνέπειε των νεοφιλελεύθερων πολιτικών η εφαρμογή αυτών των πολιτικών με τα μνημόνια, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο έχουν σαν αποτέλεσμα 25% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 28 κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση ε, ένδυας, δηλαδή 120 και παραπάνω εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν πολιτικές, οι πολιτικές αυτές έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσμα στις γυναίκες μετά από την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και μετά την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρξει αγώνας κατά της κοινωνικής ανισότητας, των διακρίσεων κατά των γυναικών και η επαναφορά ισότητας μπορεί να περάσει μονάχα με μια πολιτική κοινωνική που θα έχει εργασιακή ασφάλεια, συλλογικές συμβάσεις, αξιοπρεπή ε, αμοιβή, δημόσιες ε, ε, υπηρεσίε, οι οποίε θα είναι στον τομέα τη ε, υγείας και τη παιδεία προσβάσιμες και δωρεάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την ε, συντάκτη αυτής της έκθεσης. Είναι μια αξιόλογη και πάλι απαραίτητη έκθεση. Μας δίνει ένα σαφές μήνυμα. Οι πολιτικές λιτότητες έχουν ένα τεράστιο ολέθριο αποτέλεσμα που εκπορεύονται, μην το ξεχνάμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαν το χειρότερο αποτέλεσμα στι γυναίκε, γιατί οι γυναίκε είναι πολύ πιο ευάλωτε έναντι τη μείωση και τη κατάρριξη των δημοσίων υπηρεσιών, όπω είναι η παιδεία, η υγειονομική περίθαλψη, η δικαιοσύνη. Αυτή λοιπόν η ισότητα που θέλουμε να υποστηρίξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώ ένα αντικατοπτρισμό. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα εκατομμύρια γυναικών που είναι αντικείμενα διάκρισης και πλήττονται περισσότερο γιατί οι πολιτικές ισότητες είναι μονάχα στη θεωρία και όχι στην πραγματικότητα. Ελπίζω ότι αύριο θα υπάρξει υποστήριξη στις συστάσεις της έκθεσης της κυρίας Αρένα και θα τις λάβει επιτέλους υπόψη και η Κομισιόν. Συζητάμε απόψε την διάκριση των φύλων και την ενεργειακή φτώχεια. Μα οι κορυφαίες 7 θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν σε άντρες. Οπότε έχει λίγο δουλειά ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοπορεί π.χ. στην έρευνα και την ε, καινοτομία όπου Έχουμε βεβαίως ε, έξι μεταξύ των 25 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου και με πολλές γυναίκες. Νόμο περί ίσης αμοιβή περάσαμε το 1973 τρία χρόνια πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 52 εβδομάδες άδεια μητρότητας εγγυημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνουν τα ασφάλιστρα για γυναίκες κατά 300 λίρες το χρόνο. Τελικά για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέρος της λύσης αλλά του προβλήματος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσατε για 120 εκατομμύρια ανθρώπους ε, που ζουν σε φτώχεια. Η συγγήτρια είπε πως έχουμε 29 εκατομμύρια γυναίκες που είναι φτωχές. Άρα οι άντρες είναι οι περισσότεροι φτωχοί. Γιατί είναι λοιπόν φτωχές οι γυναίκες, γιατί δεν τις έμαθαν να είναι καλές μητέρες και σύζυγοι τους έμαθαν διάφορα άχρηστα πράγματα, αυτά περί φίλου και τέτοιες μπουρδες. Δεν έλαβε υπόψη τα στοιχεία, κύριος Κόρβιν Μίκε. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμός των γυναικών. Τα 27 εκατομμύρια που ανέφερε είναι τα παιδιά που είναι φτωχά στην Ευρώπη, λέει η κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν σκιώδης της έκθεσης αυτός, αυτής. Όμως η κυρία Ρενά και εγώ ίδια είχαμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ε, συμφωνούμε όλοι για την ε, καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας και πρέπει να πω ότι δεν καταλήξαμε στις επιθυμητές συμβαστικές λύσεις παρά την καλή μας συνεργασία. Η ομάδα μου δεν θα μπορέσει να στηρίξει την έκθεση αυτή, καθότι υπάρχουν πολλά ευαίσθητα σημεία τα οποία δεν θα έπρεπε καν να τα αγγίζει το κείμενο και δεν έχουν άμεση σχέση με τα γενεσιουργά αίτια της φτώχειας των γυναικών δεν συνάδουν ούτε καν με τις αρχές του ΕΛΚ. Αναφέρομαι όλος ιδιαίτερο στην επικουρικότητα και κάποια στοιχεία που δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μέρος της έκθεσης αυτής. Για τον λόγο αυτό δεν την στηρίζουμε, όμως θέλουμε να καταπολεμηθούν οι πηγές που προκαλούν τη φτώχεια των γυναικών. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Τόμσκι. Η κυρία Τόμσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί σειρά ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμά ή τουλάχιστον προσπαθεί να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στη δική μας πολιτική ομάδα είμαστε κατά ιασδήποτε μορφής ένδυας. Πρέπει όμως να θυμίσουμε εδώ ότι οι γυναίκες είναι ευπαθέστερες, ε, κινδυνεύουν, είναι θύματα διακριτικής μεταχείρισης και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Κάποια σημεία της έκθεσης είναι εξαιρετικά, θα τα στηρίξω. Όμως είναι απαράδεκτο σε τέτοιου είδους ψηφίσματα που είναι τόσο αναγκαία ξανά και ξανά να παρισφρίουν ιδεολογικές διεκδικήσεις. Το βρίσκω απαράδεκτο. Η αγορά εργασίας και οι σχετικές πολιτικές θα πρέπει να είναι τέτοιες που να δίδουν ε, ίσες ευκαιρίες σε όλους, ως προς την απασχόληση, ως προς τις αμοιβές, όλα τα ζητήματα. Καμία διακριτική μεταχείριση, αρνητική ή θετική, δεν είναι καλή, ούτε επιθυμητή. Εσείς μιλήσατε τόσο πολύ για την επικουρικότητα, την αρχή αυτή. Όπως είπε και ο συνάδελφος ε, πριν από μένα, δεν θα μπορέσουμε να σας στηρίξουμε στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο Επίτροπος Χίλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια, την κυρία Αρένα για την έκθεσή της σε σχέση με την ισότητα των φίλων και τις ε, επιπτώσεις ε, της διάστασης του φύλου στην Ένδια. Και είναι, την ευχαριστώ γιατί ήταν σαφής στις συστάσεις της ε, εκθεσής της. Έχει αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 64% το 2015, το γεγονό ότι έχουν χαμηλότερε αμοιβέ και υποεκπροσώψει στην αγορά εργασία οι γυναίκε. Αυτό εξακολουθεί να είναι μια πραγματικότητα, επομένω έχουν λιγότερη οικονομική ασφάλεια από του άνδρε. Όπω ακούσαμε, είναι πολύ περισσότερε γυναίκε παρά άνδρε σε ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε η κυρία Αρένα, ο κίνδυνο είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε μόνο μονογονικές οικογένειες με επικεφαλής μια γυναίκα και στις πιο ηλικιωμένες γυναίκες. Το, γεωνικό, το, το γεγονός ότι πληρώνονται λιγότερο, έχουν πολλές φορές μερική απασχόληση και κενά στην ε, απασχόλησή τους, αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις κατά 40% και πολλές γυναίκες δεν έχουν καν σύνταξη. Τον Ιούνιο του 2015 το Συμβουλίο κατέληξε σε κάποια συστήματα για το χάσμα αυτό στις ε, συντάξεις και ζήτησε να αντιμετωπιστεί στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τμήμα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τι στρατηγικές της δεσμεύσει για την ισότητα των φύλων που καθορίζουν το συνολικό πλαίσιο για τι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίε στοχεύουν να βελτιώσουν ακριβώ τη διάσταση τη ισότητα του φύλου. Οι τομεί προτεραιότητα συμπεριλαμβάνουν την αύξηση των ε, γυναικών στον χώρο τη απασχόληση, την κάλυψη του μισθολογικού συνταξιδοτικού χάσματο και το να γίνουν οι γυναίκε περισσότερο οικονομικά ανεξάρτητε. Συνεχίζουμε να δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά και προσπαθούμε να, εκδώσουμε αναχώρα στάσεις Αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα κυρίως στην έκθεσή σας αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές για την εξισορρόπηση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Πολλές γυναίκες ε, μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασία και τις χρειαζόμαστε. Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία την ε, περασμένη χρονιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξισορρόπηση αυτή και για την ε, εξέβρεση φροντιστών για άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτά είναι όλα παράδοτα για να υπάρξει ένα ευέλικτο πλαίσιο για, την, για το συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου και για υπηρεσίες ε, κοινωνικού τύπου που να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους αυτού, σε ε, όλοι οι πολίτες. Ε, σχετικές προτάσεις λοιπόν θα υποβληθούν στο τέλος της χρονιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να δημιουργήσει και έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με την ισότητα των φύλων στην καρδιά του πυλώνα αυτού. Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, αλλά έχουν οργανωθεί ευρείε διαβουλεύσει για να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασία. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη που βρίσκεται στο κέντρο της εκθέση αυτής είναι πραγματικά μια σαφής προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανένας δεν θα πρέπει να μείνει εκτός ε, της προσπάθειάς μας. Να συνεχίσουμε να προάγουμε τις προσπάθειες για την κατάκτηση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Επίτροπε για αυτά σας τα λόγια. Η συζήτηση